Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ που δείχνετε τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Καθίστε παρακαλώ για να μπορέσουμε και να αρχίσουμε. Καλωσορίζω εκ μέρους όλων των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος τα μέλη της ΙΤΡΕ για αυτή την τόσο σημαντική υπόθεση που μας αφορά και, τους, και τις δύο επιτροπές. Πρόκειται για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. Έχουμε δύο εισηγητές, τον κύριο Τούρμες, εκ μέρους της Ήτρα και την κυρία Ριβαζή, εκ μέρους της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Λυπάμαι που πρέπει να πω ότι η κυρία Ριβάση δεν τα κατάφερε να είναι εδώ, αλλά σίγουρα ο κύριος Τουρμές θα μιλήσει εκ μέρους της επίσης. Συνεπώς, Έχουμε κοινή συνεδρίαση με τον ε, συμπρόεδρο, τον κύριο Μπούζεκ, από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Πριν δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Τουρμές, θέλω να ζητήσω από τον κύριο Μπούζεκ να πει δύο λόγια για την υπόθεση αυτή. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα και από την ίδια κρίμα που η κυρία Ριβασί δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μπούζεκ, ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε όλοι μέλη της Ήτρε και μέλη της ΕΝΒΗ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική υπόθεση πράγματι. Διότι η διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ρίχνει γέφυρες με όλες τις άλλες νομοθετικές προτάσεις που έχουν να κάνουν με την Ενεργειακή Ένωση, αλλά κυρίως όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές, την ε, απόδοση κατά κάποιο τρόπο αποκτούν περισσότερη εξουσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσουμε με αυτήν την ενεργειακή μετάβαση. Από αυτή την άποψη λοιπόν πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα το οποίο ενώνει κατά κάποιο τρόπο όλες τις ε, ενεργειακές νομοθετικές προτάσεις. Στους φακέλους σας θα βρείτε και τα πρακτικά της 21ης Ιουνίου 2017. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τότε τα πρακτικά αυτά θεωρούνται κεκριμένα. Κυρία Βαλεάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θα προεδρεύσετε από κοινού με μένα. Σας δίνω και πάλι την προεδρία σε εσά για να προχωρήσουμε με τον εισηγητή. Και κυρία Βαλιάν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπούζεκ. Όπως υπόθηκε θα αρχίσουμε με τον εισηγητή, τον κύριο Τουρμές. Έχετε το λόγο κύριε Τουρμές. Για έξι λεπτά σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, δύο-τρία λεπτά χρειάζομαι μόνο και θα προσπαθήσω στο τέλος να χρησιμοποιήσω περισσότερο χρόνο. Πρέπει να σας πω ότι βρίσκομαι εδώ. Είμαι σχεδόν εκτός αιθούσης εδώ πίσω που είμαι, αλλά βλέπετε έχω παίξει ποδόσφαιρο τόσο πολύ η αγαπημένη μου θέση ήταν λίμπερο, οπότε όπως καταλαβαίνετε είμαι μια χαρά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω, όπως είπα στο τέλος, να χρησιμοποιήσω περισσότερο χρόνο, γιατί θα ήθελα να μπορέσω να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Λοιπόν, μετά από το Σαββατοκύριακο αυτό, μπορώ να πω σίγουρα και όσοι δεν μπόρεσαν να πάνε στη Φλόριντα, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι, αλλά όλο και περισσότεροι πολιτικοί ελπίζω, καταλαβαίνουν ότι το θέμα του κλίματος είναι το σήμερα. Δεν είναι τα χώαξ των Κινέζων, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, ότι πρόκειται για συνομισία ή συνομωσία που θέλει να καταστρέψει, δεν ξέρω εγώ ποια βιομηχανία. Όχι. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα αυτό τον αιώνα, το κλίμα. Πολλά έχουν γραφτεί από επιστήμονες. Και μπορώ να σας πω πώς ξεκίνησα εγώ. Το 1988 τότε στη Γερμανική Βουλή είχαμε ένα έγγραφο ε, μια επιτροπής για την κλιματική αλλαγή. Και στο έγγραφο αυτό ήδη από τότε υπήρχαν παράγραφοι που αναφέρανε την άνοδο της επιφάνειας της ε, θαλάσσης, την ε, αλλαγή της θερμοκρασίας, την αύξηση, λέει, την υπερθέρμανση του πλανήτη και έτσι σιγά σιγά αρχίζει κανείς να αλλάζει. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν είναι ένα γκώδες πρόβλημα. Δεν πρόκειται για το κατά πόσο είμαστε κοντά στο 0 το 2030 ή όχι. Το θέμα είναι πώς πάτε προς το 2050. Πάτε έτσι από πάνω ή πάτε από κάτω. Όσοι έκαναν κάποια μαθηματικά στο σχολείο, πρέπει να καταλάβουν ότι αν θέλουμε να μειώσουμε έναν όγκο, δεν μπορείτε να καθισχαστείτε από την αρχική διαδρομή. Όλοι λένε ότι ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει την επόμενη δεκαετία. Άρα πρέπει να εγκρίνουμε ένα προπολογισμό για την αντιμετώπιση του άνθρακα, να ξέρουμε τι ξοδεύουμε στην αρχή όπως κάνουμε και με τα οικονομικά μας, να κάνουμε και με τον άνθρακα. Όπως ξέρουμε τι έχουμε στην αρχή της εβδομάδα, πώς αξοδεύουμε και τι έχουμε στο τέλο το ίδιο να κάνουμε και με τον άνθρακα. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν ε, δύο πράγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν. Το ένα είναι το οικονομικό σκέλος. Εγώ προτείνω μακροπεριφερειακές συνεργασίες. Εάν, για παράδειγμα, στη Βαλτική θάλασσα. Δεν έχει σημασία αν είναι στα φιλανδικά ύδατα, στα εστονικά ή στα σουηδικά ανεμογεννήτριες, αν είναι στη θάλασσα, έτσι κι αλλιώς στην αγορά θα πέσουν όλα αυτά. Οπότε, γιατί να μην κάνουμε μια σοβαρή μελέτη για το πού είναι η καλύτερη τοποθεσία στη Βαλτική θάλασσα, μπορεί να είναι στα πολωνικά ύδατα, και να χτίσουμε με στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό φτηνά. 5.000 ξέρω εγώ πόσες ανεμογεννήτριες το χρόνο στη θάλασσα. Όλες οι χώρες να συμμετέχουν μαζί που βρίσκονται στη Βαλτική θάλασσα. Η Ρουμανία για παράδειγμα έχει φοβερό άνεμο. Έτσι πάλι στην περιφέρεια θα μπορούσε να αποφασιστεί κάτι αντίστοιχο. Αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο, συγγνώμη. Το δεύτερο τώρα. Το θέμα δεν είναι να υπάρξει συνένεση μεταξύ πολιτικών κομμάτων. Οι αλλαγές που χρειάζονται, η τεχνολογία στα κτίρια, στις μεταφορές και οι αλλαγές που χρειαζόμαστε στην οτροπία στην κοινωνία χρειάζονται τη συνένεση των πολιτών, της κοινωνίας. Είναι ψευδέστηση ότι οι κυβερνήσεις από μόνες τους μπορούν να τα καταφέρουν. Συνεπώς το δεύτερο που προτείνουμε είναι συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων, πόλεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και επιχειρήσεων. Χρειαζόμαστε δηλαδή στα εθνικά προγράμματα ένα χώρο όπου να μπορούμε να συζητήσουμε όχι μόνο ιδέες για την κλιματική αλλαγή, αλλά να συζητήσουμε πώς και ποιος θα τα βάλει όλα αυτά στο αυλάκι και θα τα εναρχιστρώσει. Ευχαριστώ και προσβλέπω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, για τον αρέα που λέγατε στη Ρουμανία, θα τα ξέρετε καλύτερα από μένα, τι να πω. Αρχίζουμε με τους σκιώδεις συζήτητες και ο πρώτος είναι ο κύριος Χόκμαρ. Γουνέρ Χόκμαν. Ευχαριστώ πολύ και επίσης να ευχαριστήσουμε και τον εισηγητή. Πρόκειται για πολύ φιλόδοξη προσπάθεια αυτή την οποία έχει τέλος πάντων καταβάλει. Και αυτό δεν είναι μόνο φιλοφρόνηση, είναι και η τοποθετησή μας. Μόνος του σχεδόν μια επιτροπή είναι. Εντάξει, αφετηρία έχουμε, τις θέσεις της Επιτροπής. Αλλά όπως και εσείς που το ποδόσφαιρο και εγώ θυμάμαι από το 1998 έχω μια άλλη εμπειρία με άλλους ε, συναδέλφους Ήμασταν στο Συνδικό Κοινοβούλιο και τότε κάναμε την πρώτη πρόταση, ούτω ώστε να υπάρχει ένα άνω όριο όσον αφορά τι εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα. Θέμα πολύ δημοφιλέ ε, τότε. Μάλλον δεν ήταν τόσο δημοφιλέ, αλλά αποσπάσαμε την πλειοψηφία. Όμως, μόνο με τη στοχοθέτηση ποτέ δεν πετυχαίνει κανείς. Θα πρέπει κανείς να προετοιμάσει το έδαφος για μηχανισμούς οι οποίοι θα φέρουν τις εξελίξεις και που εμείς ε, καταφέραμε ε, να υπάρχει ενέργεια αλλά και να ανοίξουμε την πόρτα στην βιοενέργεια και σε άλλες ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Επί τη βάση της ζήτησης προσφοράς και της καινοτομίας. Ένα κάτι που μπήκε εμβόλυμο ή καπελώθηκε πολιτικά. Υπήρχε το πλαίσιο, οπότε και είναι πολύ σημαντικό και εμείς το ίδιο να κάνουμε εδώ. Γνωρίζουμε όλοι ότι θα πρέπει να πετύχουμε τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Και όχι να κάνουμε προσεγγίρους του Τράμπα και επίσης θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, να ελοποιήσουμε αυτή την Ενεργειακή Ένωση με όλα τα θετικά της. Γι' αυτό θα πρέπει να εμείνουμε στο θέμα της διακυβέρνησης. Αυτή εδώ η έκθεση δεν είναι για χάραξη πολιτισμών, είναι για την εξασφάλιση αυτής της Ενεργειακής Ένωσης, η οποία θα αποτελεί την τήρηση των υπεσχημένων. Ένα αυτό. Το δεύτερο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να διευκολύνουμε τον ανταγωνισμό όλους που με τις ενεργικές πηγές τους μπορούν να δώσουν στους Ευρωπαίους μια ενέργεια διαφορετική, μια ενέργεια βιώσιμη, μια ενέργεια που μπορεί να εξελίξει την δημοσιογραφία της οικονομίας μας και να την προστατεύσει. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε και στα δύο μέτωπα. Το ένα δεν βγαίνει προς το άλλο. Επίσης, περιφερειακή συνεργασία εδώ θα πρέπει να επιδείξουμε προσοχή ε, και να δούμε πώ θα συγκυραστούν οι διαφορετικέ απόψει διαφορετικών κρατών μελών. Επίση, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τι διαφορετικέ αλλαγέ που αποφασίστηκαν σε σχέση με το σχεδιασμό τη αγορά, σε σχέση με την έκθεση, με την ενεργειακή αποδοτικότητα κλπ. Η διακυβέρνηση θα μας οδηγεί σε νέες πολιτικές, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι η Ενεργειακή Ένωση θα μας βοηθήσει να τηρήσουμε τις ε, υποσχέσεις μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χόκμαρ, κύριε Βαλήν, τώρα κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για την ε, ανταλλαγή που είχαμε μέχρι τώρα και ελπίζω βέβαια οι προθέσεις και οι στόχοι των συναδέλφων από τις διάφορες πολιτικές ομάδες να ληφθούν υπόψη ώστε να καταλήξουμε σε μια ευρεία συμφωνία στο Κοινοβούλιο. Η ίδια κυβέρνηση πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνει ένα εργαλείο για τον καλό συντονισμό μεταξύ του συνόλου των πολιτικών που σχετίζονται με την έρευνα και το κλίμα και για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, που θα μας δείξει το δρόμο προς τα εμπρός. Όλα τα κρατη θα πρέπει να συμμετέχουν, αλλά το κείμενο αυτό δεν θα πρέπει να είναι περιοριστικό, αλλά να είναι ένα γενικό ε, πλαίσιο για τις δράσεις που πρέπει να ακολουθούν. Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ευελιξία, γιατί αυτά έχουν τις δυνατότητες και τις γνώσεις ε, σε σχέση και με την εθνική κατάσταση για να μπορέσουν να προσαρμόσουν το ενεργειακό μείγμα καταλήλως. Σε αντάλλαγμα βέβαια τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, τηρούν τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης να έχει τα μέσα να μπορεί να επαληθεύει την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη-μέλη και συλλογικά πρέπει να φροντίσουμε να επιτευχθούν ευρωπαϊκοί στόχοι. Μία δυνατότητα, για παράδειγμα, για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. θα ήταν η χρήση ενός benchmark, ενό ε, ορίων αφοράς και κάποιων ενδεικτικών στόχων. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση αντί του να έχουμε μια εικονική γραμμική πορεία. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι η εξέλιξη δεν πάει σε ευθεία γραμμή. Σε ό,τι αφορά την εμπορική συνεργασία δεν θα σχολιάσω τα, το προλαλήσαντα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε. Πρέπει να μείνουμε ρεαλιστέ, να δώσουμε τη δυνατότητα στον καθένα να εξελίσσεται με βάση τι εθνικές ε, συνθήκες. Θέλουμε να μειώσουμε επίσης αχρία στο διοικητικό άχθο και να ενθαρρύνουμε ε, όχι όμως με στόχου, πολύ ψηλού, πολύ απομακρυσμένου από την πραγματικότητα και υπερβολικούς στόχου. Έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές ε, για τη φιλόδοξη αυτή έκθεση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει συνεργασία για μια ακόμη φορά μεταξύ Ήτρε και Ένβη. Και συνεργάζομαι με τον Κάλλο Ζωρίνιο Πιστεύω ότι οι σοσιαλιστές δίνουμε προοδευτική συμβολή σε αυτή την έκθεση. Με τους αδέλφους θα προσπαθήσουμε να καταρτήσουμε μια φιλόδοξη σχέση, έκθεση, σε σχέση με τους στόχους μας για την COP21, για να βελτιωθεί η υγεία και το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Τρεις είναι βασικοί στόχοι που επιδιώκουμε τις τροπολογίες μας κλίμα και ενέργεια, οι σχετικοί στόχοι και υποχρεώσει να συσχετιστούν μεταξύ του. Να αφαιτηθεί μια ολιστική προσέγγιση για την ενεργειακή μετάφαση και επίση να φροντίσουμε να πετύχουμε τους στόχους του 2030 και του 2050. Νομίζω αν ακολουθήσουμε και τη δουλειά που κάνει ο ΠΕΠΕ με τις ανανεώσιμες μπορούμε να είμαστε φιλόδοξοι. Η ενεργειακή παινία δυσκολεύει τις ζωές των πολιτών. Και με αυτή την έκθεση μπορούμε, έχουμε δυνατότητα να υποχρεώσουμε τα κατημέλη να αποβάλουν εκθέσει για την ενεργική παινία και να κάνουν τα απαραίτητα βήματα και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και δίκαιο ταμείο μετάβασης είναι κάτι που πρέπει να συγκροτηθεί. Είναι ευκαιρία να αλλάξουμε ε, πορεία σε ό,τι αφορά την κατανάλωση τη ενέργεια και τις συνήθειές μα. Αυτό θα αλλάξει την εργασία Βέβαια χρειάζονται στοχευμένες δεξιότητες, κατάρτιση σχετική και υποστήριξη για αυτούς που θα δουν να αλλάζουν ε, οι συνθήκες εργασίας τους λόγω ακριβώς αυτής της ενεργειακής μετάβασης. Ε, πρέπει να μας ακολουθήσουν σε αυτή την πορεία οι συμπολίτες μας. Ε, καλωσορίζω λοιπόν την προσέγγιση των εισηγητών. Άλντε και η FTD έχουν καταθέσει τροπολογίες με τις οποίες μπορούμε να συμφωνήσουμε και θα θα προσπαθήσουμε να φέρουμε κοντά μας και τις άλλες πολιτικές ομάδες με το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας. Ευχαριστώ κύριο Ζωρίνιο. Mr. Zorinio. Εκτός μικροφώνου, κύριο Ζωρίνιο, δεν τον ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, το έγγραφο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μας επιτρέπει να ευθυγραμμίσουμε την ενεργειακή με την κλιματική πολιτική. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να υπάρχει υποχρέωση να ακολουθήσουν οι χώρες μέλη. Και να διαρθρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις γύρω από τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα. Και έτσι θα έχουμε μία Ενεργειακή Ένωση, η οποία θα λειτουργεί καλύτερα και θα μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε τη δράση μας βάσει των στόχων ε, της Συμφωνίας των Παρισίων. Το βασικό έργο των εισηγητών αποτελεί μια εξαίρετη βάση εργασίας. Και έχει γίνει πρόοδο. Το είδαμε ήδη οι σκιώδεις εισηγητές μεταξύ μας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να πετύχουμε συμφωνία. Μια δυνατή συμφωνία μεταξύ των επιτροπών μας, των δύο. Αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε και σημαντική πλειοψηφία στην Ολομέλεια όταν ψηφίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι πέρα από την ευθυγράμμιση αυτή των δύο ενιών ενέργεια και κλίμα, όπως γίνεται στην έκθεση αυτή, μιλάμε και για βιωσιμότητα. προκειμένου να πετύχει η ενεργειακή μετάβαση, να μην υπάρχει ανισότητα απέναντι στην ενέργεια. Μιλάμε για μέσα παραγωγής, ανάπτυξη. Να λοιπόν γιατί πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σαν βάση αυτό το έγγραφο, εμείς οι δύο επιτροπές, για να κινητοποιήσουμε και τους υπόλοιπους συναδέρφους ώστε να υποστηρίξουν και εκείνοι και να καταλήξουμε σε μια δυνατή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια. Στο τέλος των διαπραγματεύσεων είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε μια πλήρη έκθεση με συνοχή που να σέβεται τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Πρέπει επίσης να δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και αυτό σημαντικό. Η έκθεση αυτή πρέπει να στεφθεί από επιτυχία. Και εμείς, όπως το είπαν θα είμαστε ανοιχτοί στην πολιτική μας ομάδα, ώστε όλοι μαζί, όλες οι πολιτικές ομάδες, να φροντίσουμε να επιτεθούν οι κοινοί μας στόχοι. Ευχαριστούμε πολύ καλή αυτή η δήλωσή σας. Ο κύριος Στοσανόφσκι έχει τώρα το λόγο. Θα σας μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα, στα τσεχικά. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Το έργο τους είναι πάρα πολύ εξαιρετικό και οι προτάσεις τους. Βέβαια τα πράγματα με τίποτα δεν είναι απλά, πρέπει να τα συζητήσουμε κι άλλο και θέλω κι εγώ να σταθώ σε αυτό που μας είπε ο Κλόντ προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τι οικονομικέ παραμέτρου στην έκθεση, διότι δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζουμε μόνο κάποια ιδεολογήματα και όλα αυτά να μην είναι με οικονομικό τρόπο αποτιμητά. Θα πρέπει να δούμε ποιε θα είναι οι συνέπειε για την οικονομία του κάθε κράτου μέλου επίση. Ε, θέλω να έρθω και να συμφωνήσω και με τον Κουναρχόρμα και με τους άλλους συναδέλφους που ανέφεραν ότι όντως είναι πάρα πολύ βασικό το κάθε κρατός μέλος να έχει κίνητρο από αυτήν την έκθεση. Να μην θεωρηθεί μόνο μια αγκαρία διοικητική το πώς θα συμπληρωθούν τα έντυπα, τα κουτάκια, οι πίνακες θα πρέπει να έχουν κίνητρο τα κρατημέλη και έτσι να φροντίσουν για το μέλλον έχουμε συμφωνήσουμε αυτό που άκουσα επομένω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κρατημέλη να είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις με ευελιξία και να υπάρχει έτσι ένα περιθώριο Άλλες συνθήκες επικρατούν σε κάθε κράτος. Αλλού είπαμε ότι υπάρχει άνεμος που βοηθάει πάρα πολύ, ε, αλλού υπάρχει κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό. Επομένως, θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε και την περιβαρική συνεργασία. Ήδη έχει αρχίσει γιατί είναι κάτι το που μας ξεπερνάει, κάτι πολύ μεγάλο αυτές οι μεταβολές στον ενεργειακό μέτωπο. Αλλά θα πρέπει τι γίνεται με τα συστήματα μετάδοσης, ε, με τις ανταλλαγές των κρατών μελών και να μην παραφορτώσουμε γραφειοκρατικά τους μηχανισμούς ελέγχου. Γιατί έτσι θα σκοτώσουμε την τόσο σημαντική έρευνα. Για τον κόσμο πολύ σημαντικό να μπορεί να έχει φθηνή ενέργεια. Το τελευταίο που θέλουν οι Ευρωπαίοι είναι κάποια αρχή να τους λέει ότι έχει το όριο του 1,5% κλπ. κλπ. Εντάξει, να έχεις ένα στόχο, ας πούμε, το 1,5% αλλά δεν προχωράει έτσι η τεχνολογία. Μπορεί για μια χρονιά το 1,5% να γίνει 4,5%. Γι' αυτό και ελπίζω ότι τελικά θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια λογική λύση. Κύριε Μπούζεκ, ευχαριστώ για το ότι προείδρευσε στο πρώτο ήμιση της συνεδρίασης. Έχουμε 1.500 τροπολογίες. Τρομερή δραστηριότητα από όλους τους συναδέλφους. όπως και οι συγκητές μας βέβαια για όσες τροπολογίες φτιάξαμε. Πάμε τώρα στους επόμενους από τους σκιώδες ηγητές που έχουν ζητήσει το λόγο. Πάντως κάποιοι από τους εκείνους ε, είναι στην Ολομέλεια, θα έρθουν αργότερα, επομένως δεν μπορούμε να τηρήσουμε την προβλεπόμενη σειρά. Οπότε από τους σκιώδες ηγητές έχουμε εδώ τους εκπροσώπους του EFTD. Τον συνάδελφο Νταρίο να από την Ήτρα. Έχετε το λόγο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Η διακυβέρνηση της Ενεργικής Ένωσης είναι ένα μεγάλο όραμα, ένας πολύ σπουδαίος στόχος που έχουμε τάξει η προς το παρόν 28. Και η ενέργεια είναι το θεμέλιο του τι θα κάνουμε για την κλιματική αλλαγή. Έχουμε δει όλες αυτές τις εικόνες ε, της ισοπαίδωσης, πρώτα στο Τέξας, μετά στο Μαϊάμι της Φλόριντα, ε, αλλά ε, και υπάρχουν και άλλες τέτοιες θεομηνίες στο Μαγκλαντές, στη Σχήρα Λεόνια, δεν είναι τόσο γνωστές. Ακόμα και εμείς έχουμε στην Τοσκάνη και στο Λάτιο πλημμύρες. Και εγώ, και εγώ έχω συναδέλφους που τους πλημμύρισε το σπίτι και επίσης ε, είχαμε και πνιγμούς κάποιων ε, παιδιών. Οπότε έχουμε ιστορική ευθύνη να έχουμε ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο όπως επίσης και για τις ανέμενες πηγές ενέργειας και για την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα να υπάρξει επομένως στο ύψος των περιστάσεων μια διακυβέρνηση στο ύψος των συμφωνιών του Παρισιού και να μην κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Να τηρούμε τα, τα υπεσχημένα, να μην κάνουμε όπως κάποιοι άλλοι μεγάλοι κάνουν. Οπότε αυτή, ε, αυτό, το, αυτό το σχέδιο κανονισμού ε, αφορά όλο, μια ολόκληρη μέτρων, αλλά θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη. Εμείς συμφωνούμε και με τους δύο εισηγητές ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. 40% για το ανανεώσιμο, 45% όσον αφορά την ενεργειακή. Α, όχι αντίστροφα διορθώνει, 45% ανανεώσιμο, 40% η ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι ιστορική αυτή η βάση που ζούμε. Και Ε, θα πρέπει να προσέξουμε όπως σε όλες τις κρίσιμε περιόδους αν θα γκρεμίσουμε ή θα χτίσουμε αυτό που έχουμε. Και είπαμε λοιπόν, για την παράγοντο οικονομία αλλά είδατε η οικονομία πώς καταστρέφεται από αυτές τις θεομηνίες. Ούτε επιχείρησεις μπορούν πρέπει να λειτουργήσουν γιατί όλα ε, υφίσταται αυτή την απερίμωση όπως και η γεωργία. Μα τι θα φάμε, τι θα φάνε τα παιδιά μας, τι μέλλον θα προετοιμάσουμε για τον πλανήτη. Δεν είναι θέμα οικονομίας, είναι θέμα ύπαρξης της ανθρωπότητας. Αυτό διακυβεύεται για την προσπάθεια για σταθεροποίηση του κλίματος. Συμφωνούμε με τους εισηγητές. Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο χρειάζεται και έτσι όλοι να εμπλακούν σε αυτές τις προσπάθειες για τις ανέφημε πηγές ενέργειας και για την ενέργεια με κοινωνικό πρόσωπο και όχι να στηρίζεται μόνο στην αγορά γιατί η αγορά δεν είναι πάντα η θέση του να κυβερνήσει μια οικονομία ή μια ήπειρο ή έναν πλανήτη ολόκληρο. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για τις παρατηρήσεις σας. Επόμενος και ο δίσπαος του κατάλογό μου ε, είναι πρόσωπος του ΙΕΝΕΦ. και συγκεκριμένη συνάδελφος κυρία Μιρέγη Τορνανό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιέπαινο είναι να θέλουμε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα φαινός και να κάνουμε πιο ασφαλή τον ενεργειακό εφοδιασμό αφετέρου. Ωστόσο, η Ένωση Ενεργειακή που θα επιβάλλει δεσμευτικούς στόχους στο σύνολο των κρατών μελών δεν είναι κάτι που μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Δεν ε, είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σας πενθυμίσω ότι με βάση τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία καθορίζουν από μόνα τους ε, το ενεργειακό τους μείγμα. Επομένως δεν έχει καμία αρμοδιότητα και δεν μπορεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργειακή μετάβαση ως κάτι καταναγκαστικό διότι έτσι θα ήταν σοβαρές καταστροφικές οικονομικές και κοινωνικές απώλειες για πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες που συνεχίζουν να εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα σε μεγάλο βαθμό. Για τις περιοχές αυτές όμως η Κομισιόν δεν προβλέπει κανένα σχέδιο βιώσιμης αναδιάρθρωσης δεν είχε λύσεις η Κομισιόν μακροπρόθεσμα να προσφέρει ό,τι αφορά την ενεργειακή αυτάρκεια. Είναι ένας ευσεβής πόθος μόνο. Αυτός λοιπόν ο Ναβουχοδονός από τον Ναμπούκο, το... ο αγωγός αυτός είναι η πανάκια που είχαν βρει και τελικά εστέφθη με μια μεγάλη, ήταν πάρα πολύ αποτυχημένο ως project. Θέλει τώρα να δημιου... η Κομισιόν να δημιουργήσει την Ενεργειακή Ένωση, όμως ε, δεν έχει ορίσει ούτε τα πλαίσια ούτε τη... τους στόχους. Το θέμα είναι να σεβαστούμε τι αρμοδιότητες των κρατών μελών, όπως προβλέπεται από τις συνθήκες. Ευχαριστώ. Thank you very much, madame. ευχαριστώ. Γκερμπράντι, Κονέτσνα, Πετριτσίνη. Φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι αυτοί θα έρθουν με κάποια καθυστέρηση ίσως, γιατί εξακολουθούν στην Ολομέλεια. Να περάσουμε λοιπόν σε άλλους ομιλητές. Η ε, κυρία Κροστέτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν ήδη. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το κείμενο αυτό για τη διακυβέρνηση είναι κεντρική σημασία. Γιατί είναι αυτό που θα αποτελέσει τη σύνδεση ανάμεσα στα διάφορα κείμενα για την ενέργεια που εξετάζουμε αυτή την εποχή. Πρέπει όμως να παραμείνει ένα γενικό πλαίσιο. Γιατί πρέπει να επιτρέψει να παραμείνει ευελιξία στις χώρες μέλη. Η εμπειρία που έχω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσα πολλά χρόνια που είμαι, ε, μου δείχνει ότι οι οδηγίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικέ από τις χώρες μέλη, καταλήγουν να γίνουν μια τρύπα στο νερό. Σύμφωνα, σύμφωνα υπάρχει η Συμφωνία των Παρισίων και πρέπει να τη σεβαστούμε. Όμως κάθε χώρα μέλος πρέπει να μπορέσει να υποφεληθεί από αυτή την ευελιξία και να αποφασίσει από μόνη της η κάθε χώρα την κατεύθυνση που θα πάρει για να σεβαστεί ακριβώς τις δεσμεύσεις μας απέναντι στη Συμφωνία των ε, Παρισίων. Οι χώρες μέλη λοιπόν πρέπει να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους βάσει των διάφορων ε, τεχνολογιών. Θα πούνε τι θα προωθήσουν περισσότερο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους. Γιατί το ενεργειακό πρόβλημα δεν είναι πάντα το ίδιο σε όλες τις χώρες. Οπότε πρέπει οι χώρες να έχουν ε, την διευκόλυνση αυτή να αποφασίσουν για τον ενεργειακό τους μείγμα. Είναι επίσης ενδιαφέρον στα εθνικά σχέδια να αναλύουμε και τις συνέπειες των εθνικών μέτρων που θα ληφθούν ε, για την τιμή του άνθρακα για παράδειγμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να ευνοήσουμε επενδύσεις και να επιτρέψουμε και στους επενδυτές να βλέπουν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Οπότε ναι, να είμαστε απαιτητικοί να τηρηθούν οι συμφωνίες των Παρισίων, αλλά να αφήσουμε ευελιξία στις χώρες μέλη, απαιτώντας συγχρόνως από αυτές να πάρουν τις καλές αποφάσεις και αυτές τις αποφάσεις να τις αναλύουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Πιλάρδη Δικαστήριο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γιατί υπόθηκαν ήδη πολλά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν πτυχές όπως είναι η ευελιξία που έρχονται και επανέρχονται. Γιατί είμαστε τελικά πολλοί εκείνοι που πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η ευελιξία ε, στο γενικό πλαίσιο. Όσον αφορά το άρθρο 4 εφόσον στόχος μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, για να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει κάθε χώρα μέλος να μπορεί να συνεισφέρει με ευελιξία για να μπορέσει να επικεντρωθεί σε αυτό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα στην κάθε χώρα. Με άλλα λόγια δηλαδή, να μην ξεχνάμε ότι στην κάθε χώρα υπάρχει διαφορετική πορεία για τις ανανεώσιμες, και οτιδήποτε άλλο διάφορες τεχνολογίες σε διαφορετικό βαθμό χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες. Κάτι άλλο τώρα για την ε, ενή αγορά ενέργειας. Από τις 28, δύο δεν έχουν καν πετύχει την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο όπως θέλουμε. Δηλαδή μπορεί τελικά να παραμείνει κάτι σαν ευσεβής πόθη όλο αυτό που λέμε για την συνδημότητα. Λοιπόν, πρώτον, να λάβουμε υπόψη μας τα εθνικά προγράμματα και την πορεία της κάθε χώρας όσον αφορά την ηλεκτρική συνδεσιμότητα. Δεύτερον, να προτείνουμε οι χώρες μέλη να πούνε πώς θα πετύχουν τους συγκεκριμένους στόχους και η Επιτροπή να αξιολογεί βάσει αυτού τα εθνικά προγράμματα και τέλος οι χώρες που δεν έχουν αρκετή διασυνδεσιμότητα να φροντίσουν να προχωρήσουν στις ανανεώσιμες πηγές ανάλογα με το βαθμό διασυνδεσιμότητας και να, λάβουν, να λάβουμε υπόψη μας την, ε, το μειωμένο αυτό βαθμό διασυνδεσιμότητας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιαβόρν, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπαν οι συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θέλω όμως να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, θέλω να σας υπενθυμίσω το αποτέλεσμα μια άλλη υπόθεσης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, όπου η ΕΝΒΗ συμφώνησε με μια ιδιαίτερα φιλόδοξη γνωμοδότηση όσον αφορά την οδηγία αυτή. Να ενισχύσει το στόχο σε 40% για το 2030, δεσμευτικά κτλ. Και πολύ μου αρέσει το αποτέλεσμα, αλλά όλες αυτές οι φιλοδοξίες θα γίνουν πραγματικότητα μόνο αν έχουμε και ένα σημαντικό πρόγραμμα διακυβέρνησης για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ακριβώς αυτούς τους στόχους στο πακέτο καθαρής ενέργειας. Άρα χρειάζεται ένα θεματικό και δυνατό πρόγραμμα ενεργειακής διακυβέρνησης για να πετύχουμε τόσα αναφέρουν οι άλλες οδηγίες όπως για παράδειγμα εκείνη της ενεργειακής απόδοσης, εκείνη για τις ανανεώσιμες κλπ. Δεύτερη παρατήρηση. Θα ήθελα να τονίσουμε ιδιαίτερα την βοήθεια για τα νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων. Και το άρθρο 19 και το άρθρο 29 στο κείμενο που εξετάζουμε πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο για να ενισχυθούν τα πιο φτωχά νοικοκυριά ε, στην Ευρώπη, πιο φτωχά απέναντι στην ενέργεια. Και γι' αυτό ζητάω τα άρθρα αυτά 19 και 29 να ενισχυθούν ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες αυτούς που δεν έχουν αρκετή πρόσβαση στην ενέργεια, γιατί δεν πρόκειται μόνο για τις ανανεώσιμες, στην ε, ενεργειακή απόδοση κτλ. Πρόκειται και γι' αυτό, για να μπορούν όλα τα νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση στην ενέργεια. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Κόρβιν Μίκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τους ε, συναδέλφους ε, των Πρασίνων και τι είπανε για την υπερθρέμψη του πλανήτη και σκέφτηκα τι γίνεται με αυτές τις μία αλήθειες, με τις ειδήσεις, ειδήσει, με την αλλίωση της ε, αλήθειας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά είναι θέματα για ψυχίατρο, αλλά όμως ε, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι στην ηγεσία της Ευρώπης βρίσκονται κάποιοι με φιλοδοξίες πολιτικές και εδώ και πολύ καιρό έχουν φτάσει και έχουν βγει στην Ευρώπη σε μηδενική ανάπτυξη. Και όλες τους ενέργειες εκεί κατατείνουν στο να έχουμε μηδενική ανάπτυξη. Οπότε όλα αυτά τα μία λυθή αυτό εξυπηρετούν αυτό το στόχο τη μηδενική ανάπτυξη. Ευχαριστούμε για όσα μα είπατε, λέει ο πρόεδρο και τώρα, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κονέτσνα, η οποία είναι η σκιώδη συζητητρία για την Ευρωπαϊκή Νοτική Αριστερά. a Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη που άργησα. Ήταν πολύ σημαντική η συζήτηση στην ε, Ολομέλεια και άλλωστε ήταν κάτι που σχετιζόταν με το θέμα μας. Τέλος πάντων συμπαθάτε με που άργησα. Τον Ιούνιο στην κοινή μας συνεδρίαση είπαμε ότι ελπίζουμε πως αυτή η έκθεση θα τύχει συζήτησης ε, ευρεία και ελπίζω ότι έτσι θα γίνει πριν φτάσουμε στην ε, ψηφοφορία του Νοεμβρίου θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με όλη αυτή τη δεσμή μέτρων και ο τίτλος αυτό υποδηλώνει ότι όλοι θα πρέπει να καλυφθούν και πρέπει να δούμε πώ θα υπάρξουν κάποια μέτρα αποτελεσματικά και από πλευρά ε, κόστου, Όπου δεν ισχύει κάτι τέτοιο, οι προτάσει είναι λάθος. Και μην έχουμε επικάλυψη επίσης των ε, επιμέρους πολιτικών του καθενός. Όταν λέμε εδώ για νέο ETS, αυτές οι τροπολίες που στο ETS, σε τι ακριβώς αναφέρονται. Οι συνάδελφοι του που τις ε, υπέβαλαν αυτές οι τροπολογίες. Αναφέρεται στο και το θέμα τη ε, επικάλυψη. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα όρια τη ευθύνη εκάστου και το σύστημα λίγης των εκπομπών ETS και οι ευθύνε τέλο πάντων που αναλογούν στον καθένα. Και θα πρέπει να δούμε ποιος αναλαμβάνει ποιο κομμάτι τη ε, προβληπόμενη πολιτική. Έχουμε 500 τροπολογίες. Έχουμε και κάποιες φιλόδοξε, οπότε θα πρέπει και το Συμβούλιο να ξέρει πώς έχουν τα πράγματα στη δική μας ζήτηση. Έχουμε ήδη προσπαθήσει να καταλήξουμε σε συμφωνία. Η πολιτική μας ομάδα δεν ενθουσιάστηκε πραγματικά βλέποντας την έκθεση Πίπερ. Πάντως όσοι την εγκρίνατε να μην ξεχνάτε ότι οι προτάσεις για ενεργειακή αποτελεσματικότητα αν εγκριθούν θα οδηγήσουν σε συρρήγνωση των τιμών για το σύστημα ETS. Ε θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό το σύστημα. Έτσι. Θα υπάρξει κατάχρηση των μέτρων και άρα αυτό αντιβαίνει στους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξιδίου. Χρειάζεται περισσότερη μείωση των εκπομπών. Θα σταματήσει η πολιτική περιορισμού τη του άνθρακα να είναι αποτελεσματική όλοι θα υποστούμε τις συνέπειες. Άρα ας εναρμονίσουμε τις πολιτικές των κρατών μελών. Ας εναρμονίσουμε τα των μέτρα. Ας πάμε όλοι μαζί στο κοινό στόχο, δηλαδή τη μείωση του άνθρακα. Επίσης να εναρμονιστούν και οι στόχοι που έχει θέσει ο καθένας και όλοι φυσικά να τηρήσουν τους στόχους που έχουν τεθεί. Πείτε, Λίζε, επόμενος. Ο κύριος Λίζε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ ζητώ συγγνώμη καταρχάς γιατί άργησα να φτάσω επειδή ταυτόχρονα στην Ολομέλεια υπήρχε η συζήτηση για τις εκπομπές από την αέρα κυκλοφορία. Κατά την άποψή μου και στα δύο θέματα, αυτό δηλαδή που συζητήθηκε στην Ολομέλεια και αυτό που συζητούμε εμείς τώρα εδώ, η προστασία του κλίματος, η Συμφωνία των Παρισίων είναι στο πρώτο πλάνο, είναι στην πρώτη γραμμή και σε ό,τι αφορά την προστασία του κλίματος, ε, ε τραγικά επίκαιρο το θέμα, όπως είδαμε και βλέπουμε ακόμη στις ειδήσει ε, των τελευταίων ημερών. Αυτά που γίνονται τώρα στην Νότια Ασία, στην Καραϊβική, στις ΗΠΑ, αυξάνουν και σε οξύτητα και σε συχνότητα και θα συνεχιστεί να γίνεται αυτό αν δεν κάνουμε κάτι για την καταπολέμηση αλλαγής του κλίματος και αυτό για μένα είναι το σημαντικότερο γιατί θέλουμε απαλλαγή από άνθρακα με αυτή την έκθεση. Αυτός είναι ο βασικός στόχος ε, και σίγουρα ε, για τη δική μου πολιτική ομάδα, όπως άλλοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ουδέτερη τεχνολογία, ανοιχτή τεχνολογία. Σίγουρα και η παραγωγή ρεύματο είναι σημαντικό. Έχουμε στόχους από την Κομισιόν που πρέπει όμως να συγκεκριμενοποιηθούν σε ό,τι αφορά ε, το ρεύμα, σε ό,τι αφορά την ε, ε, απαλλαγή από τον άνθρακα. Σε άλλους τομείς βέβαια είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και το έχουν συζητήσει και στην ομάδα των 7 στο G7 σε ό,τι αφορά τους στόχους της βιομηχανίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διακυβέρνηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη σχετική προσέγγιση, θα μπορούσε κανείς να το συζητήσει διαμακρών. Ο Γιάβορ επίσης ε, μίλησε για την ενεργειακή απόδοση 40%. Το ΕΛΚ την προηγούμενη εβδομάδα καταψήφισε αυτή την πρόταση θα μπορούσαμε να επιχειρηματολογήσουμε για αυτό το ποσοστό, ε, αλλά ε, το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε σε άλλες συμβαστικές προτάσεις ε, σε ό,τι αφορά παραδείγματο χάρη τους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους, τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αν δεν μπορούμε να το πετύχουμε με δεσμευτικούς εθνικούς Ευρωπαϊκού, να δούμε τι θα γίνει με του εθνικού στόχου. Και έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις για αυτά τα όρια αναφορά στα benchmarks και να μπορούμε να συζητήσουμε κατά πόσον αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας κυρίες συνάδελφε και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα είναι εδώ η κυρία Ρίτσαρτς, Διευθύντρια της ΓΔ Ενέργεια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετέχουμε, να ακούσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες τις παρουσιάσεις. Ε, πραγματικά θαυμάζω τη φιλοδοξία που θέλησε να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρόταση αυτή και αναγνωρίζουμε ότι αυτό είναι μια πολύ θετική πτυχή. Από την άλλη πλευρά θεωρούμε ότι οι στόχοι που σχετίζονται με τους διάφορους τομείς θα πρέπει να παραμείνουν σε τομεακή νομοθεσία. Σε ό,τι διαφορά τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του όλου πακέτου, αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ σημαντικό και θυμάμαι στην τελευταία συνάντηση, την τελευταία κοινή συνεδρία στον Επιτροπή Ιτρέμβη και εσείς κύριε Μπούζα και κυρία Βαλεάν επενθυμίσατε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση, συνολική προσέγγιση για το πακέτο αυτό. Ήθελα να αναφέρω και κάτι ακόμη, συγκεκριμένα ότι το όλο αυτό πακέτο συνάδει απόλυτα με την ενεργειακή μετάβαση στην αλλαγή του κλίματος, αλλά είναι και μια ευκαιρία για μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερε θέσει εργασία. Άρα καμία σχέση με μηδέν ε, ανάπτυξη. Θα να το τονίσω αυτό. Θέλω να φέρω και κάτι άλλο γενικό, ότι δηλαδή αυτό που ελπίζαμε είναι να κινηθούμε με ταχύς ρυθμούς για να δώσουμε το μήνυμα και στον υπόλοιπο κόσμο ότι είμαστε σοβαροί προ που αναλάβαμε στο πλαίσιο τη Συμφωνία των Παρισίων και θέλουμε να προχωρήσουμε τάχιστα προ τα εμπρό. Σεβόμαστε βέβαια και λαμβάνουμε υπόψη τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας απόψεις. Θέλω τώρα να περάσω σε κάποια πιο συγκεκριμένα σχόλια και επιτυχές. Πρόκειται για έναν τομέα όπου ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση θα λάβει υπόψη τις συλλογικές, ε, ε, τα συλλογικά επιτεύγματα και τους στόχους του 2030. Μεταξύ άλλων θέλουμε να έχουμε ε, ως δυνατόν νωρίτερα συμφωνία με τους άλλους εισηγητές. Είπα ότι πρέπει να είναι συνεκτικό και συνεπές συνολικά αυτό το, το πακέτο. Αναγνωρίζουμε ότι είναι ουδέτερο να υπάρχει ουδετερότητα σε εθνικό επίπεδο. Εσείς μιλάτε για δεσμευτικούς εθνικούς στόχους, αυτό είναι ενδιαφέρον, είναι φιλόδοξο όμως και πρέπει να το συζητήσουμε. Και εσείς πρώτα απ' όλα να το συζητήσετε για το των τα σχέδια εθνικών προγραμμάτων. Υπάρχει μια προθεσμία που είναι σημαντικό να τηρηθεί για να μπορέσουν να δοθούν και επενδυτικά μηνύματα. Γιατί κάποιοι μιλήσατε για ότι είναι, ότι είναι σημαντικό, είπατε, να δοθούν ε, μηνύματα προ την αγορά για επενδύσει. Και ο διάλογο είναι σημαντικό στο πλαίσιο τη Συμφωνία των Παρισίων. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο, θα παραμείνει ψηλά ο πύχη ό,τι αφορά τη φιλοδοξία αυτή τη πρόταση. Εκτιμούμε ιδιαίτερο τη στήριξη που προσφέρεται στην περιφερειακή συνεργασία, γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πώς να το πω. Αυτό που θα ήθελα να πω ως προειδοποίηση, μην είμαστε τόσο περιοριστικοί και να μην κατονομάζουμε περιφέρειες. Ξέρουμε ότι ο ενεργειακό τομέα έχει αλλάξει δραματικά. Μόνο τα τελευταία 10-15 χρόνια να δείτε. Μπορεί να είχαμε μία περιοχή για το ρεύμα Χ και μία περιοχή για φυσικό αέριο Ψ. Αλλά αλλάζουν αυτά και πρέπει να βρούμε τι πιο καλέ λύσει. και δεν πρέπει να είμαστε άκρο περιοριστικοί, μειώντα τα σύνορα, τα όρια κάποιων περιοχών. Σίγουρα η περιφερειακή συνεργασία είναι απαραίτητη και οι διασυνδέσει μεταξύ των κρατών μελών θα προωθήσουν την νέα ενεργειακή αγορά και θα βελτιώσουν τι εμπορικέ μα σχέσει με άλλε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση Έχετε λοιπόν καταθέσει πολύ ενδιαφέρουσες, πολλά υποσχόμενες τροπολογίες. Θα τις ε, μελετήσουμε και θα τις συζητήσουμε μαζί σας, ε, βέβαια πάντοτε έχοντας υπόψη και τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στο Συμβούλιο. Μια άλλη πτυχή που κάποια από εσάς αναφέρατε και την οποία και εμείς θεωρούμε σημαντική είναι η ενεργειακή παινία και η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα στο μέλλον. Αν με επιτρέπετε όμως τώρα θα ήθελα επειδή έφυγε ο συνάδελφος από το Γενική Διεύθυνση Κλίμα, να διαβάσω τη σημειώση που μου άφησε, αν μπορείτε να σταματήσετε το χρονόμετρο. Ωραία, λοιπόν, άρα, ε, πολλές σημειώσεις εδώ που μου είχε αφήσει πρόσωπος, θα, θα περιοριστώ σε κάποια. Θέλουμε να ενισχύσουμε μία συγκεκριμένη πτυχή που έχει να κάνει με τη μακροχρόνια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιος από τους στόχους του 2050 προτείνεται κάποιες από τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει. Ναι, μεν εκτιμούμε τη φιλοδοξία, αλλά είναι λίγο πρόωρο κατά την άποψή μας να το εντάξουμε στο πλαίσιο του κανονισμού για τη διακυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το συνδυασμό πολιτικών και μέτρων μεταξύ ETS και ενεργειακής απόδοσης, σημειώνουμε την ανησυχία σας σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα του ETS. Στόχος κοινό είναι αυτός, αλλά θεωρούμε ότι το θεματικό ή τη σταθερότητα της αγοράς που πρέπει να ισχύσει ε, από το 2019 θα ανταποκριθεί στις ανάγκες ανεξαρτήτως οικονομικών παραγόντων και εξελίξεων. Σε ό,τι αφορά τις ε, προθεσμίες για την υποβολή αναφορών και το στόχο να μην υπάρξει για τα κράτη-μέλη πρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος, και εδώ εντάσσονται και τα εθνικά σχέδια. Σε κάποιες προθεσμίες είμαστε λίγο πιο αυστηροί στον κανονισμό διακυβέρνησης ε, σε σχέση με το MMR, αλλά αυτό το κάναμε για να υπάρξει ένας εξορθολογισμός και τα κράτη-μέλη να μπορούν να αντιδρούν και να συνεργάζονται από κοινού. Ο εκπρόσωπο τη Δέλτα Κλίμα μιλά για την Επιτροπή για την Αλληλεγγύη του κλίματο, την Επιτροπή Μύφιν, για τη σχέση μεταξύ κλίματο και χρήση γη, Επειδή όμω δεν σχολιάστηκαν αυτέ οι πτυχέ, ίσω θα ήταν καλύτερο να σα τα υποβάλουμε γραπτός όταν θα συζητούμε τι μεμονωμένε τροπολογίε. Ευχαριστώ. Πούτζεκ, ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε. Τώρα, οι συγγητέ μα, Δηλαδή ο Κλόντ Τούρμας, γιατί η κυρία Μισελ Ριβασί είπαμε δεν είναι μαζί μας. Κλόντ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιους ε, από εσάς, ίσως όχι όλους. Ο κύριος Σόκμαρ έχει δίκαιο όταν λέει ότι οι αγορές πρέπει να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Σε ένα κόσμο που έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανώσιμες πηγές ενέργειας, δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί, κανένας υπάλληλο που να μπορεί να τις διαχειριστεί. Είναι οι αγορές. Όμως, Κουτμαρ, όταν λες ότι η επιτυχημένη σουηδική πολιτική βασίζεται σε μια αγορά πράσινου πιστοποιητικού, αυτή δημιουργήθηκε από τους πολιτικούς στη Σουηδία. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να θέσει ένα στόχο. Και η αγορά αυτή είναι εντελώς ε, τεχνητή, αλλά αναγκαία με το πράσινο πιστοποιητικό. Άρα πρώτα είναι η πολιτική η οποία καθορίζει τις αγορές αυτές. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Άρα χρειαζόμαστε στόχους. Το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τις υποδομές. Μπορείτε να έχετε, και ο κύριος Κανιέτε γι' αυτό, τις καλύτερες προθέσεις ε, για την κινητικότητα με ηλεκτρικά οχήματα, αλλά αν δεν υπάρχουν σταθμοί φόρτισης, ο κόσμος δεν θα αγοράσει. Ή μπορείτε να, έχετε, να θέλετε να έχετε μια εξαίρετη offshore εγκατάσταση ε, ανεμογεννητριών, αλλά πρέπει να υπάρχει σύνδεση. Υπάρχει το καλώδιο, αλλά πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερο σχεδιασμό όπως ίσως γινόταν σε κάποιες κομμουνιστικές χώρες. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα όραμα και μετά να βάλουμε το μείγμα των υποδομών και των αγορών. Δεύτερον, κυρία Ντελέη, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό και αυτό είναι η συγκρισιμότητα ανάμεσα στα διάφορα εθνικά σχέδια. Είπατε ότι μπορούμε εύκολα να επαληθεύσουμε. Μα πώς θα επαληθεύσετε τα σχέδια του 2050 αν δεν έχετε προηγουμένως κανένα κριτήριο. Η μια χώρα θα στείλει μια μισή σελίδα, η άλλη χώρα θα στείλει 150 σελίδες. Οπότε η μόνη τροπολογία που έκανα με την Ιδρύ και με άλλους είναι να έχουμε στόχο τη συγκρισιμότητα. Δηλαδή να φτιάξουμε μισή σελίδα κριτηρίων όχι για να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά για να διασφαλίσουμε την ύπαρξη της συγκρισιμότητας. Για τις ανανεώσιμες, η ελάχιστη πορεία, λυπάμαι, αλλά ίσως θα πρέπει να σας δώσουμε μια σύνοψη του τι γίνεται στο Συμβούλιο. Οι χώρες μέλη είναι υπέρ της ε, πορείας αυτής τελικά, γιατί πρόκειται για την ασφάλεια επενδύσεων. Η ιδέα αυτή ότι οι χώρες ενδεικτικά θα πούνε τι ίσως θα κάνουν χωρίς να έχουμε καμία λεπτομέρεια για να ξέρουμε κατά πόσο ακολουθεί την ε, προκαθορισμένη πορεία ή όχι το κράτος, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει βεβαιότητα έτσι για επενδύσεις. Τερέσα Κρίφιν, αγωνίζεστε για την ε, έλλειψη αποκλεισμών. Και έχετε δίκιο. Θα υπάρξουν τομείς της οικονομίας όπου θα χάσουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε στη βιομηχανία ότι ο άνθρακας έχει μέλλον. Όχι, τελείωσε ο άνθρακας. Αλλά αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στον άνθρακα. Να μην είναι αυτοί οι χαμένοι. Αυτό ναι. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επόμενο έγγραφο για την Ενεργειακή Ένωση θα έρθει όχι μόνο με χρήμα, αλλά και με ιδέες. Το πρόβλημα της αναδιάρθρωσης μιας περιοχής που βασίζεται στον άνθρακα δεν είναι μόνο το οικονομικό. Πρέπει να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες. Και μια περιφέρεια που εφαρμόζει μια λάθος πολιτική δεν μας βοηθάει πολύ όσο μια άλλη η οποία έχει επιτυχία. Συνεπώς, χρειάζεται πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε ναι, να υπάρξουν και χρήματα για αυτές τις περιοχές που θα κλείσουν ε, οι μονάδες άνθρακα, αλλά να έχει και ιδέες τι θα γίνει με τους εργαζόμενους εκεί. Εδώ προσπαθούμε να πετύχουμε μια συνένεση γύρω από αυτή την ιδέα. Η ενεργειακή παινία έχει να κάνει με την πρόσβαση σε χρήματα. Αν δεν έχω χρήματα, δεν μπορώ να είμαι συνδρομητή σε κάποιο δίκτυο, δεν μπορώ να πληρώσω για τη μόνωση του σπιτιού μου, οπότε ναι, πρέπει να καταπολεμηθεί αυτή η ενεργειακή παινία. Ναι, κύριε Ζωρίνιο, πρόκειται για το Παρίσι, όντως. Το θέμα είναι πώς θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο Παρίσι. Και μια από τις ιδέες που εισάγουμε είναι ότι το Παρίσι έρχεται με πενταετής κύκλους. Και γι' αυτό και η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να ακολουθήσει. Και όπως προσπάθησα να εξηγήσω και την προηγούμενη φορά, αυτό θα ενισχύσει και την ασφάλεια επενδύσεων, τη βεβαιότητα. Κύριε Ζωνενόφσκι, έχετε δίκιο. Πρόκειται για την οικονομική επάρκεια. Ναι, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ανατολική Ευρώπη. Έχετε δύο είδων προβλήματα. Γιατί μια ανεμογεννήτρια στην Ρουμανία κοστίζει 10-15 φορές παραπάνω, ενώ η ίδια ανεμογεννήτρια στη Γερμανία έχει 3%. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και γι' αυτό λέω ότι θέλω λύσεις, ώστε να μπορούμε να έχουμε χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειωθεί το κόστος στη Ρουμανία, στην Ελλάδα, στην Πολωνία. Και το δεύτερο είναι τι κάνουμε με χώρες όπως η Σλοβεν... όχι η Σλοβενία μάλλον, η Σλοβακία, η Τσεχία, το Λουξεμβούργο εύκολη πρόσβαση σε αυτούς που έχουν offshore εγκαταστάσεις. Δεύτερες χώρες δεν έχουν θάλασσα. Με 5.000 ΜΒ. Γιατί να μην μπορεί να ανοίξει ο διαγωνισμός, να είναι 60% για τη Δανία ή 40% για την ή 10% για την Τσεχία, 10% για το Λουξεμβούργο, 10% για τη Σλοβακία. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο και στην Ελλάδα, την Ισπανία για την ηλιακή ενέργεια. Χρειάζεται αλληλεγγύη δηλαδή μεταξύ των χωρών μελών. Για να φτάσουμε εκεί όμως χρειάζεται διάλογο σε πολιτικό επίπεδο. Και γι' αυτό και προτείνω εταιρικέ σχέσεις μεταξύ των χωρών μελών. Ένα από τα προβλήματά μας στην Ενεργειακή Ένωση είναι ακριβώς το ένας ή 28 μαζί. Αλλά αυτό δεν βοηθάει να υπάρξει εμπιστοσύνη. Α βάλουμε τις βαλτικέ χώρες μαζί για να δούμε τι θα κάνουν στη βαλτική θάλασσα. Εμπιστοσύνη μπορεί να σημαίνει χώρες γύρω από τη Μεσόγειο, μπορεί να σημαίνει η Πιλάρ. Και θα τελειώσω με αυτό. Πολύ τυχερός είσαι γιατί έχουμε χρόνο. Αλλά στο μέλλον θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα λεπτό. Μα ως εισηγητής πρέπει να έχω παραπάνω, λέει ο κύριος Τι Πιλάρ, εγώ προτείνω Ισπανία, Πορτογαλία και η Ιταλία μαζί να μπουν στο κλαμπ. Αν θέλετε περισσότερες σχέσεις με τη Γαλλία, προτείνω Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία που αποτελούν μέρος αυτού του πόλου να δουλέψουν μαζί η Αυστρία, η Γερμανία και η Γαλλία ενδεχομένω σε άλλα σχέδια για εκεί. Θα σταματήσω εδώ. Και ευχαριστώ για την υπομονή σας συνάδελφοι που με ακούσατε. Μπούζε, σε σταμάτησα Κλώτ και με συγχωρείς. Έχουμε ακόμη 13 λεπτά. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ συνάδελφοι. Όπως γνωρίζετε καλά, ο συντονισμός είναι πάρα πολύ αναγκαίος για αυτή τη δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια. Είναι βέβαια κυρίως αρμοδία η Ήτρε, αλλά έχουμε συνεργαστεί για αυτό το θέμα και έχουμε 1500 τροπολογίες, έχουμε και τις συμβαστικές, όλα από τις τραπέζες είναι αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας και ο συνήθως ο Κλοντ εξαερώνεται. Ο εκθάμενος εξαφανίζεται αμέσως μετά την ομιλία του. Σπάνιος, σπάνιος βουλευτής. Δεν είναι, εμείς τον έχουμε, εσείς δεν τον έχετε στην ένδυ τέτοιον βουλευτή. Δύσκολο να βρείτε τέτοιον βουλευτή. Κι όμως τα άκουσα όλα όσα είπες και σε ευχαριστώ, λέει ο Κλοντ. Α, Πολύ σημαντικό. Το τελευταίο μήνυμα από πλευρά μου. Στις 28 Νοεμβρίου έχουμε την ψηφοφορία. 5 η ώρα. 28 Νοεμβρίου, 5 η ώρα. Φέτος, πολύ σημαντικό. Απαραίτητη η παρουσία σας. Το δε. Δεν θα έχουμε και άλλα, άλλα δύο θέματα. Πέντε ώρα. Το πρωί θα συνεδριάσει Ήτρε, αλλά Ήτρε με ενβία. Εκείνη συνεδρία στο απόγευμα. Βαλέα Ας έχουμε ξεκάθαρο μυαλό να μην μπερδεύουμε και άλλο αυτό το θέμα, ε, να καταλήγουμε σε μια αξιολογική πρόταση από την Επιτροπή και εύχομαι όλοι πάρα πολύ επικοδομητικά να συμβάλλετε. Καλό βράδυ, ευχαριστώ και τον Πρόεδρο Μπούση.